9 η ώρα το πρωί. Έχει δημοσιευθεί και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του διαδικτύου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το ημερήσια διάταξη και